Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε λίγο καθυστερήσει, αλλά θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να τηρήσουμε το ωράριό μας. Όπως ε, έχετε καταλάβει, διαβάζοντας το πρόγραμμα ήδη, είμαστε εδώ σε μια συνάντηση που πηγαίνει πέρα από την δημοσιονομική πειθαρχία. Πώς να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσης απασχόλησης και την κοινωνική πρόοδο κάτω από οικονομικές συνθήκες οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές. Είναι τιμή μας που έχουμε μαζί μας δύο επιτρόπους και θα τους δώσω βεβαίως τον ε, λόγο σε λίγο. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι, που είναι εκείνο ο οποίος χειρίζεται ακριβώς τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και έχουμε και τον Επίτροπο Χάν, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει με ιδέες σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές και τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων, ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τις περιφέρειές μας και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του για να δούμε ακριβώς πώς τα θέματα της ανισότητας ή της ανάγκης για ανάπτυξη, επενδύσεων κτλ. πώς μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά, όπως επίσης και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, πώς θα ενταχθούν στον επόμενο προγραμματισμό. Ο πρόεδρος Φαναρομπάη το είπε πριν στην Ολομέλη, αλλά επιμένω και εγώ και το επαναλαμβάνω ότι ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τους προπολογισμούς των κρατών μελών, τελικά χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο για πράγματα όμως τα οποία φαίνεται ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ο Φαντουροπά είπε ότι είναι ένας προϋπολογισμός καταρχήν επενδυτικός. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά πάντως εκείνος είναι πεπισμένος και αποφασισμένος για μια κλίδα ε, κατανομής μεταξύ των χωρών και Επίσης, πρέπει να σας πω εδώ ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν κινητοποιείται ένας προπολογισμό σε επίπεδο χώρας μέλου. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό στην άσκηση αυτή 2012 για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να βάλουμε να συνεργαστούν και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Απασχόλησης. Γιατί αυτό το οποίο σήμερα ζητάνε οι Βρυξέλλες εντό εισαγωγικών από τις χώρες μέλη για τους προπολογισμού τους, γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο χρέωσης των χωρών μελών, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα όσον αφορά τις απενδύσεις. Κοιτάμε λοιπόν την χρέωση, αλλά όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μιλάμε καθόλου για την χρέωση αυτή. Ενώ μέσα στη λιτότητα και τη σοβαρότητα που πρέπει να έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία, η κινητοποίησή μας γύρω από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι διαφορετική από εκείνη στα πλαίσια των χωρών μελών. Θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Όμως, πέρα από αυτά που είπαμε στην Ολομέλη, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι για την προσπάθεια που κάνουμε μεταξύ μας. Διότι εδώ και χρόνια τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Συζητιούνται προτάσεις για τη δημιουργία, τα διαβάζω αυτά εδώ και εκεί, ε, νέων σωμάτων. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το οποίο είναι το καθήκον μας ως ευρωβουλευτές, τον, κοινο, τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο του προπολογισμού, για παράδειγμα. Πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας, να έχουμε διασκέψεις διακοινοβουλευτικές, υπάρχουν τέτοιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι, αλλά και ο καθένας στο δικό του το επίπεδο να ασκεί πλήρως τον κοινοβουλευτικό του ρόλο. Είτε εμεί εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κινητοποιούμεθα για να λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που πιστεύουμε εμείς για την ανάπτυξη, και ξέρετε τι έχουμε αποφασίσει και όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και όσον αφορά την απασχόληση. Και από την άλλη μεριά εσείς να κάνετε επίσης τη δουλειά σας σε εθνικό επίπεδο για να δείτε σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται με τον προπολογισμό και πώς αυτός ενορχιστρώνεται. Χωρίς άλλη καθυστέρηση όμως θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι για να μας εισάγει στη συζήτηση και μετά θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Τεχάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκλησή σας. Ειλικρινά νιώθω ακόμα σας στο σπίτι μου εδώ. Ξέρετε ότι ήμουν στην Επιτροπή Προπολογισμών εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι' αυτό το λέω αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι όταν κάνουμε τη σύγκριση αυτή, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε κανεί όντω να βρει τι διαφορέ. Το ένα είναι το θέμα του ελλείμματος είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, το θέμα των πολιετών επίσης προγραμμάτων που καλύπτει πολλές φορές. Και επίσης το ότι είναι επενδυτικό. Ξέρω το επίπεδο επενδύσεων στο, στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, Πολωνία, που είναι 5%. Άρα μπορεί κανείς εύκολα να δει τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη σαν επένδυση αλλά αυτό ακριβώ είναι που συζητιέται τώρα. Πώ με τα χρήματα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση και πώ να έχουμε ε, καλό ανταγωνισμό, ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη τι χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει μια νέα ιστορία να διηγηθεί για να ξεπεράσουμε τους σκεπτικισμούς. Δεν μπορεί να είναι η παλιά ιστορία που λέγαμε, που είχε να κάνει με την ειρήνη, γιατί δεν είναι τα πράγματα τα ίδια σήμερα όπως ήταν τότε. Εδώ χρειάζεται να παγιωθεί η δύναμη της Ευρώπης και να μην θεωρείται αυτό σαν πρόκληση σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στα πλεονεκτήματα που μας ενώνουν και να να καταδείξουμε ότι εμείς έχουμε τα εργαλεία για την λύση. Μπορούμε ή δεν μπορούμε. Αυτή θα ήταν μια καλή ιστορία για να ε, μπορεί να διηγηθεί η Ευρώπη και όχι τις παλιές τη Περιδίνης κλπ. Επίσης, χαίρομαι που βλέπω μια πιο ισορροπημένη πρόταση για ένα οικονομικό μείγμα πολύ περισσότερο σήμερα από ότι το 2009 και το 2010 γιατί τότε η λιτότητα ήταν ε, η μητέρα κάθε πολιτικής δεν σκεφτόμασταν ε, τίποτα άλλο τώρα η προσέγγιση μας είναι πολύ πιο ισορροπημένη προσπαθούμε να έχουμε ανάπτυξη επενδύσεις και φορολογικά μέτρα επίσης υπέρ της ανάπτυξης. Δεν φτάνει βέβαια η φορολογία. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε και τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι γίνεται με την ανεργία των νέων, που είναι η χαμένη γενιά της Ευρώπης. Αλλά ακριβώ έτσι πρέπει να τοποθετούμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μέσα στα πλαίσια αυτού του οικονομικού μείγματο εν μέσω κλίματος λιτότητας. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό αποτελεί μια πραγματική εργαλειοθήκη, στην οποία μέσα έχουμε και το μαστίγιο και το καρότο. Το μαστίγιο χρησιμοποιήθηκε ε, κατά της Ουγγαρίας ε, όχι ε, υπήρχε μια παύση, μια άρση που κρατάει μέχρι του χρόνου. Και υπάρχουν κι άλλα όμως μαστίγια που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Όμως μέσα σε αυτή την εργαλειοθήκη έχουμε και το καρότο που δεν έχει να κάνει μόνο με την διευκόλυνση, την οικονομική, αλλά έχει επεκταθεί και περισσότερο και στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Η διευκόλυνση των ε, πληρωμών επίσης και εκτός Ευρωζώνης για την Λετωνία και την Ρουμανία. Τώρα αποτελεί μέρος του πακέτου διάσωσης για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όμως, πάνω από όλα αυτά, και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη φύση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, το βασικό λοιπόν είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία ως μέσον προώθησης με πολλαπλασ... ως πολλαπλασιαστικό φαινόμενο δηλαδή διάφορα προγράμματα. Έχουμε 8 χώρες με πολύ ψηλή ενέργεια των νέων, Σλοβακία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία. Όλες αυτές οι χώρες είναι ανοιχτές και αυτό είναι το μήνυμα, πιστεύω, που θα έρθει και από τον συνάδελφό μου, τον Γιωχάνης Χάν, σε λίγο. Αχ, αυτό θυμάμαι σαν καλό από το κοινοβούλιο σε σχέση με εμά ότι εδώ προσφέρεται καφέ και τσάι. Λοιπόν, συνεχίζω, λέει ο κύριος Λεβαντόφσκι είμαστε πια ε, ανοιχτοί και ετοιμαζόμαστε για τον ε, επαναπρογραμματισμό των διευθυντικών ταμείων. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Είμαστε έτοιμοι. Είναι κάτι που έχει γίνει για τις χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και πάνω απ' όλα η Ελλάδα με υψηλό συντελεστή συγχρηματοδότησης, δηλαδή 10% παραπάνω δίνει η Ευρώπη από το δικό της προϋπολογισμό και μόνο 5% έρχεται τελικά από την ενδιαφερόμενη χώρα. Εμεί δηλαδή συν 10% φτάνουμε στο 95% και 5% οι χώρες. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια μεγάλη ανακούφιση στις μέρες μας. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μπορώ να παριθμίσω διάφορα, αλλά θα το κάνει νομίζω ο Γιωχάνες που θα σας εξηγήσει πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω πρόσβασης σε μικροπιστώσεις. Πρέπει να δοκιμάσουμε και την ιδιωτική αγορά βέβαια μέσω επενδυτικών ομολόγων που δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε με γιατί ο όρος αυτός ε, εκνευρίζει ορισμένους. Θέλουμε λοιπόν να δοκιμάσουμε τη ιδιωτική αγορά μέσω τέτοιων επενδυτικών ομολόγων στο μέλλον. Έτσι πιστεύω ότι θα καλύψουμε ένα κενό στην χρηματοδότηση, τη διαφορετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να στηρίξουμε έναν καλό προϋπολογισμό, 1% του ΑΕΠ, λιγότερο δηλαδή από ό,τι είχαμε ανάμεσα στο 93 και το 99 που ήταν 1,8 του ΕΠ τώρα ανάμεσα στο 2000 και το 2013 είναι 1,06. Και φροντίζουμε εξάντε να υπάρξει πάγωμα στον προπολογισμό μέχρι το 2020 με 1% στις πληρωμές. Διαθέτει λοιπόν τα εργαλεία του προπολογισμού αυτός. Φροντίζουμε για μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, δηλαδή αυτό το οικονομικό μείγμα στην Ευρώπη, Άρα έχουμε πραγματικά εργαλεία για να ενισχύσουμε την απασχόληση αλλά και να διατηρήσουμε από την άλλη μεριά τις ε, αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη. Μίλησα 7 λεπτά, αλλά ναι, εντάξει, ήταν κάπως εκτενής η εισαγωγή μου. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς να καθυστερώ, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Χάν να μην ξεπεράσουμε στον χρόνο του κύριου Λεβαντόφσκη, ώστε και οι βουλευτέ να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η πολιτική συνοχή είναι πολιτική ανάπτυξης το ιστορικό καθήκον της πολιτικής συνοχής ε, ήταν να δημιουργήσει μια σύγκληση μεταξύ των ε, ανισορροπιών που υπήρχαν μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Αυτή είναι σήμερα και, αυτό είναι σήμερα και το κεντρικό της ε, καθήκον, να προωθήσει την πολιτική ανάπτυξη, οι αδύναμες δηλαδή οι περιοχές να γίνουν πιο ισχυρές, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ισορροπία με τις υπόλοιπες πιο δυνατές περιοχές. Η περιφερειακή λοιπόν πολιτική, η πολιτική συνοχή ήταν πάντα πολιτική ανάπτυξη και ειλικρινώς σας λέω ότι θα ήθελα να μιλούμε για ε, ταμεία ανάπτυξης αντί για ταμεία συνοχής και ταμεία διαρθωτικά, γιατί τα δύο τελευταία, τα τελευταία ακούγονται πολύ ε, γραφειοκρατικά. Με το Ταμείο Ανάπτυξης περιγράφουμε αυτό ακριβώς που, αυτό ακριβώς που θέλουμε να πούμε. Θα ήθελα την εισαγωγή μου να τη μοιράσω σε δύο μέρη. Να σας πω καταρχάς ε, το τι κάνουμε τώρα ή τι έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Γιατί πολλές φορές ε, υπάρχει έτσι μια κατηγορία ότι η διαρθρωτική πολιτική, δηλαδή η πολιτική ανάπτυξης, δεν είναι παρκώς ευέλικτη. Είμαστε ευέλικτοι γιατί ακριβώς αποκινούμε τα κράτη-μέλη, είμαστε σε θέση όταν υπάρχουν ε, πρωτοβουλίες να, που μπορούμε να τις υποστηρίξουμε δηλαδή από τα κρατη να ε, ε, προσαρμόζουμε τα διάφορα λειτουργικά προγράμματα και να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι τα διάφορα λειτουργικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία τώρα εκπονούνται ουσιαστικά έτυχαν διαπραγμάτευση το 2005-2006. Τότε ο κόσμος είχε τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι έχει σήμερα. Οπότε προφανώς πρέπει τώρα να απαντήσουμε. Για να απαντήσουμε λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα. Και το θέμα δεν είναι απλώς να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, είναι να πούμε ότι ναι, τώρα πρέπει να απαντήσουμε με ανάπτυξη. Προφανώς όλοι περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα και βέβαια πρέπει να δούμε ποια είναι και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε. Τους τελευταίους 12 μήνες, στα πλαίσια και του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, έχουμε 345 προγράμματα. 161 ε, προγράμματα, περίπου δηλαδή τα μισά, τροποποιήθηκαν. 6,3 ε, δις ευρώ εισέρευσαν ναι, ε, επιπλέον, όσο επιπλέον κονδύλια προς τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών. Και αυτό έγινε ε, σε 20 από τα 27 κρατημέλη. Επίσης, απαντήσαμε στην κρίση γιατί ήδη από το 2009 και το 2010 αυξήσαμε τις προκαταβολές και έφτασε αυτό το ποσό περίπου στα 7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ μπήκανε στην αγορά για να υπάρξει α, α, χρήμα καινούριο και να κινηθεί η αγορά. Το προηγούμενο έτος είχαμε επίσης αυξήσει τους δείκτες χρηματοδότησης μέχρι το 95% σε μερικές περιπτώσεις. Βεβαίως αυτό οδήγησε στο να υπάρξει περίπου ένα δισεκατομμύριο ε, ευρώ το οποίο να πάει ε, σε κράτη για, τις, για τα επιχειρησιακά τους ε, προγράμματα. Επίσης, τα revolving funds Επίσης θα ενισχύσαμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε διάφορες αγορές, όπου ας πούμε το κλίμα για, τις, για την πίστοση των, ή για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν πολύ άσχημο. Έχουμε λοιπόν και αυτό το επιχειρησιακό κεφάλαιο πια. Προσπαθούμε και από κοινού βεβαίω με τα κοινοβούλια σας αλλά και με το Συμβούλιο να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια, ένα εργαλείο ε, κατανομής κινδύνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τα διάφορα προγράμματα που υπάρχουν, ακριβώς επειδή υπάρχει και η σχετική πρωτοβουλία του Προέδρου Μπαρόσο για τις 8 χώρες οι οποίες πλήττονται σοβαρά από την ανεργία των νέων. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εκεί και πώς μπορούμε να ε, αλλάξουμε λίγο την κατανομή των, ε, των κονδυλίων έτσι ώστε να μπορέσουμε στοχοθετημένα να στείλουμε αυτά ακριβώ τα κονδύλια στι ε, επιχειρήσει που πλήττονται. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που έχουν γίνει. Βεβαίω αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Πώ δηλαδή τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Αν τώρα δούμε γενικώ πώς έχει η κατάσταση, ε, με εκπλήσει πρέπει να σας πω το γεγονός ότι για το κοινωνικό ταμείο το ποσοστό απορρόφησης είναι αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με το περιφερειακό ταμείο και νομίζω ότι ακριβώς σε, τόσες, ε, σε τόσο δύσκολες ε, καταστάσεις για την, ε, για την αγορά θα πρέπει και το ταμείο αυτό να χρησιμοποιηθεί και ειδικώ από τις χώρες που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Γιατί πραγματικά απορώ πώς γίνεται να μην χρησιμοποιούνται οι, οι δυνατότητες που δίνονται και που διατίθενται στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη συζήτηση που γίνεται και χαίρομαι πολύ που μπορούμε να την κάνουμε σήμερα εδώ. Βεβαίω, πρέπει να εξελιχθούν κι άλλο τα πράγματα και αυτό είναι και το αντικείμενο της διάσκεψης αυτής. Ε, πρέπει επίσης να πω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ε, μία, έναν οδικό χάρτη σύγκλησης για την Ευρώπη. 12, ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων την προηγούμενη εβδομάδα σε μια, έστειλαν μια επιστολή στον, στον πρόεδρο Μπαρόσο και στον πρόεδρο Φαν Ρομπάι ε, για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, την ολοκλήρωση της ε, ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, ήταν μερικά από τα αιτήματα σε αυτή την επιστολή. Όλοι, αυτό, όλοι αυτοί είναι τομεί όπου εμεί δραστηριοποιούμεθα, αλλά βεβαίω όπου τα κράτη-μέλη, από τα κράτη-μέλη μάλλον, ζητείται να κάνουν και να δώσουν και αυτά την συμβολή του. Και όταν μιλούμε για συμβολή, δεν μιλούμε μόνο για χρήματα, μιλούμε και για πολιτικέ αποφάσει. γιατί, εκεί, γιατί μονίμως γίνεται μια συζήτηση για αυτό. Ε, εν συντομία λοιπόν αυτά ήταν κάποια σημεία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο και να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλύτερα τα εργαλεία που έχουμε, σύμφωνα βεβαίω και με τα αποτελέσματα που έχουν δώσει ήδη. Γιατί το να ε, στοχοθετήσουμε το πρόγραμμα μα ανάλογα με τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε και θεματικέ προτεραιότητε. Και σα το λέω ε, με τα λόγου γνώσεω αυτό. Αυτέ οι προτεραιότητε. πρέπει να τεθούν. Ε, Βεβαίω, όταν ε, υπάρχουν ε, προτεραιότητε, μονίμω έχουμε ένα πρόβλημα με το ποιε θα είναι οι προποθέσει που θα πρέπει να πληρούνται. Έχουμε 11 προτεραιότητε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλέ δυνατότητε. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, κύριε Επίτροπε, για να μπορέσουμε να θέσουν και ερωτήσει και να λάβουν και απαντήσει οι βουλευτέ. Δύο λεπτά και θα, θα σιωπήσω για το υπόλοιπο της συνεδρίασης, αν θέλετε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω, προτείνουμε ε, είμαστε ε, ε, έχουμε θέσει ως στόχο μας ε, τα αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε και την ε, προπόθεση της αιρεσιμότητας για να δούμε κατά πόσο μπορούν όλες αυτές οι προτεραιότητες να ε, λειτουργήσουν. Και βεβαίως αν θέλετε ευχαρίστω να σας απαντήσω σε σχόλια ή ερωτήσεις εάν έχετε. Αυτοί όμως είναι οι βασικοί πυλώνες αυτής της αρχιτεκτονικής και πρέπει να διατηρηθούν έτσι ώστε οι πολιτικές να είναι πιο ορατές, πιο απτές και πιο αξιόπιστες για τους Ευρωπαίους πολίτε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Θα είμαι πολύ λιγότερο ανεκτική με τους βουλευτές, κανονικό είναι αυτό. Να δώσω το λόγο καταρχάς στο Λάζλο Σοριάν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του δώσω το λόγο για ένα τρίλεπτο. Merci beaucoup, hogy ε, három perc azt jelenti, hogy magyarul fogok beszélni. Az Európai Unió fantasztikus Τρία λεπτά μου είπατε να μιλήσω. Ε, με ρίξατε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε 20 ε, έχουμε 20 εκατομμύρια λιγότερους φτωχούς, όπως λένε οι δείκτες. Ε, οι δείκτες όμως ε, στο σύνολό τους έχουν χειροτερεύσει. Για να λύσουμε λοιπόν τα κοινωνικά προβλήματα χρειάζονται λεφτά. Όταν όμω 18, χρο... 18 χώρες έχουν πολύ ψηλά ε, ελλείμματα, τότε προφανώς τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη που δεν ε, τα έχουν πάει τόσο καλά θα πρέπει να μάθουν το μάθημά τους και να δουν ποιο είναι το μυστικό των χωρών που τα έχουν πάει καλά. Ε, μία δυνατότητα θα ήταν ε, τα κονδύλια της Ένωσης ε, να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Φέτος μιλούμε για 82 δισεκατομμύρια. Μέχρι το τέλος του 2011 χρησιμοποιήθηκαν το, το μισά από αυτά. Προφανώ πρέπει το πράγμα αυτό να αλλάξει. Η Κομισιόνα έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, ε, έδωσε τι προκαταβολέ, έκανε πιο γρήγορα τι πληρωμέ. Επίσης ε, ε, ε, ενίσχυσε τον δίκτυ χρηματοδότηση. επομένως πρέπει και τα κράτη-μέλη από τη δική τους τη μεριά να προσπαθήσουν να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους απορρόφησης αυτών των κονδυλίων. Οι στόχοι λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες της κρίσης. Η Κομισιόν το είπε, αλλά δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες. Θα πρέπει να δούμε γιατί η παραγωγή ε, φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επανεγκαθίστανται αλλού οι ε, επιχειρήσει. Βεβαίω αυτό είναι δική του υπόθεση, δεν μπορούμε να του εμποδίσουμε, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να ε, δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Υπάρχουν ναι χώρε που έχουν χαμηλότερου μισθού, αλλά η μοντέρνα σκλαβιά που κρύβεται σε αυτέ τι χώρε και μιλώ για την παιδική εργασία πρέπει να, το, πρέπει να τη δούμε, να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μάλιστα νομοθετικά. Ε, επίσης, ε, να δούμε τι γίνεται με τους ε, κανόνες για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος κτλ. Βεβαίω όλα αυτά καθιστούν την εργασία ή την παραγωγή πολύ πιο ακριβή και βεβαίω οι εταιρείε πηγαίνουν σε χώρε όπου δεν χρειάζεται να πληρούν όλε αυτέ τι προποθέσει. Το θέμα όμω είναι ότι το ΑΕΠ τη Ένωση με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και οι εισαγωγές πιέζουν πάρα πολύ την παραγωγή των κρατών μελών. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, καθώς επίσης και την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος. Γιατί ας πούμε δεν υπάρχει οικολογικός φόρος. Ε, Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να σημάνουμε συναγερμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αναλύσουμε σοβαρά την κατάσταση και εγώ προσπάθησα να το κάνω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι που μα δώσατε μια εικόνα τη κατευθύνσεω που θα ακολουθήσετε. Σαν συγκεκριτή τη Επιτροπή Προπολογισμών, ονόμα τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κορνέλισεν, που ήταν η συγγήτριά μα όσον αφορά την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την ετήσια εξέταση τη ανάπτυξη. Έχετε στα έγγραφά σα το ψήφισμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα της εκθέσεως που συνετάχθη. Η κυρία Κορνέλησεν έχει για ένα τρίλεπτο το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, καλώς ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό εμείς σαν και από τις δύο πλευρές να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο διότι θέλουμε να είναι ένας δρόμος προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη. Θέλουμε να δείξουμε πόσο αλληλένδετες είναι οι οικονομίες μας. Ε, εγώ είμαι υπέρομαχος των στόχων του 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διότι θεωρητικά όλα αυτά θα λειτουργούσαν υπέροχα. Τα κράτη-μέλη θα έθεταν τους στόχους, θα συνέτασαν συγκεκριμένα προγράμματα για να κατευθυνθούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση και τελικά το 2020 να έχουμε πετύχει του στόχου μα. Η υψηλή απασχολησιμότητα, χαμηλά επίπεδα φτώχεια, πολλή καινοτομία, υψηλά επίπεδα παιδεία. Δεν είναι ανέφικτα όλα αυτά. Στην πράξη όμω αυτά δεν λειτουργούν τόσο καλά. Οι καινοί στόχοι περσινοί ήταν μονόπλευροι και αυτό το λιγότερο μπορώ να πω. Αγνοώντα τι κοινωνικέ πτυχέ και την ανεργία. Πολλέ χώρε δεν κατέβαλαν προσπάθειε να εφαρμόσουν εθνικά μεταρρυθμικά προγράμματα κατεύθυνση προ το μέλλον, απλώς ε, αναμόρφωσα κάποια προγράμματα που ήδη είχαν. Πρέπει να ομολογήσω ότι το πρόβλημα τη Ολλανδία, τη χώρα μου, ήταν ένα αρκετά απογοητευτικό και καταθλιπτικό παράδειγμα αυτού. Αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν έχει ακροατήριο. Οι βουλευτές ε, δεν συμμετέχουν πολύ, ελάχιστα, οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμμετέχουν, η κοινωνία των πολιτών δεν συμμετέχει, ε, ο τύπος δεν συμμετέχει, οπότε δεν ελέγχονται λοιπόν οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν ε, κάκιστα εθνικά προγράμματα. Ε, έχω κάποιο μήνυμα για τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν συζητείτε το πρόγραμμα της χώρας για την ε, μεταρρύθμιση στα κοινοβούλια σας, σκεφτείτε τα εξή. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά πρώτα απ' όλα. Η χώρα σας, το, πρόγραμμα της χώρας σας είναι ένα τμήμα ενός συνόλου των 27 χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ισχυρό σύνολο να αντιμετωπίσει την κρίση και να βγει ισχυρότερη από την κρίση αλλά μόνο αν όλοι επενδύσουμε σε μια καινοτόμα οικονομία με το ανάλογο εργατικό δυναμικό. Οι χώρες που μπορούν θα πρέπει να επενδύσουν στην κοινή μας οικονομία, ώστε να αφαιρηθούν όλοι. Ενώ οι χώρες που θα πρέπει να τακτοποιήσουν τους προϋπολογισμούς θα πρέπει να το κάνουν. Θα πρέπει να δείτε, επενδύει 3% στην καινοτομία χώρα σας, επενδύει αρκετά στην παιδεία. Δεύτερο, σκεφτείτε μακροπρόθεσμα. Τα εθνικά προγράμματα, τα μεταρρυθμιστικά, τα φετινά, είναι τα δεύτερα σε σειρά από τα δέκα. Θα πρέπει να κοιτάζουν προς το μέλλον. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το μέλλον είναι η γυράσκουσα κοινωνία. Σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλές κενές θέσεις σε πολλές χώρες και θα χρειαστούμε όποιον μπορεί να εργαστεί, να εργαστεί από την αγορά εργασία. Επενδύει αρκετά στους νέους η χώρα σας προετοιμάζει τους νέους για τη γύρανση των κοινωνιών. Η χώρα σας επενδύει σε μέτρα για την συν... να συνδυάζεται ο χώρος εργασίας με την μέρημνα, με την πρόνοια για να συμμετέχουν οι γυναίκες. Σχεζόμαστε. Χρειάζεται συνεχτική προσέγγιση. Ένα από τα βασικά προβλήματα σε πολλές χώρες είναι και το εξής τα σχέδια είναι προφανώ σύνδετα, δεν έχουν συνοχή. Αν από τη μία πλευρά λένε οι κυβερνήσει θέλουν να μειώσουν τη φτώχεια και από την άλλη πλευρά κάνουν περικοπέ όσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα, τι συντάξει και τα μέτρα για την ενίσχυση τη αγορά τη εργασία, Άρα δεν θα πετύχουν τελικά το στόχο τη πιθανότητα. Αν λένε από τη μία κυβερνήσει ότι θα προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και από την άλλη ε, δεν υποστηρίζουν τη μέρημα των παιδιών, πιθανότατα δεν θα μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή των ε, γυναικών στην αγορά εργασία. Μετά θα πρέπει να σκεφτείτε δημοκρατικά. Θα πρέπει εσείς να γίνετε οι ακροατές ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εμείς το ίδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα σα. Η αντιπρόεδρο τώρα τη Επιτροπή για την Εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση του Κυπριακού Κοινοβουλίου που αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομα, η κυρία Σκέβη Κούντρα Κουμά. Η σημαντικότητα του ρόλου των κοινοβουλίων στη συζήτηση για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης εγκείται κυρίως στο γεγονός ότι τα κοινοβούλια ως εκπρόσωποι του λαού μπορούν και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές που θα χαράσσονται θα είναι ανθρωποκεντρικές θα πρέπει να είναι οι εκφραστέ τη ε, θέση ότι θέματα όπω η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και κεκτημένων των εργαζομένων που απειλούνται από το λεγόμενο νοικοκύρεμα των προπολογισμών, θα πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχετική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών οι επιπτώσει τη παγκόσμια οικονομική κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία καθώ και η συνεπακόλουθη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη, είχαν άκρο αρνητική επίδραση στον τομέα της απασχόλησης. συμμερίζομαι τι ανησυχίε που έχουν διατυπωθεί από διάφορε κατευθύνσεις σε σχέση με τι αποφάσει που έχουν ληφθεί τον περασμένο δεκέμβριο. πρόκειται για αλλαγέ που στο όνομα της νομισματικής σταθερότητας οδηγούν σε περαιτέρω εκχώρηση της κρατικής κυριαρχίας των μελών της ένωσης ενώ η ρήτρα για μόνιμα ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση των κοινωνικών πολιτικών διολίσθηση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων αύξηση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών όξιση της ανεργίας και ειδικά της νεανικής και γυναικείας. η δημοσιονομική πειθαρχία και νομισματική αυστηρότητα δεν πρέπει να αποτελεί σκοπό αλλά ένα εργαλείο στην πρόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Περαιτέρω επίκεντρο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση των θέσεων εργασίας. Οι προϋπολογισμοί σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίνουν έμφαση στι δημόσιε επενδύσει, όπω την έρευνα, την καινοτομία. Έχουν ακουστεί αρκετά σήμερα και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Πιστεύω όμω ότι χρειάζεται ένα καινούριο σχεδιασμό για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών τη κρίση, τη ανεργία, τη αυξανόμενη φτώχεια, τη έλλειψη αναπτυξιακή όθηση προ παραγωγικού τομεί των οικονομιών. Θα ήθελα δηλαδή Χρειάζεται ακόμα ένα νέο σύμφωνο εργασίας και ανάπτυξης που θα επιτρέπει στα κράτη να ακολουθούν ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που ισχύουν σε κάθε χώρα και σίγουρα όχι αποτέλεσμα επιβολής άλλων ισχυρών κρατών ή των μονομερών επιταγών της αγοράς και του συστήματος. Θα ήθελα δηλαδή να δω την Ήπειρο μας μια ενωμένη Ευρώπη που θα ελέγχει τα κράτη-μέλη της όχι αν ευημερούν οι αριθμοί, αλλά κατά πόσον πετυχαίνουν να μειώνουν την ανεργία, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες, να διασφαλίζουν δημόσια δωρεάν και ποιοτική παιδεία και υγεία για τους λαούς και να τιμωρεί τις κυβερνήσεις όταν δεν τα πετυχαίνουν αυτά. Δηλαδή ένας ριζικός αναπροσανατολισμός του δρόμου κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθείται στην Ήπειρο μας βέβαια όταν μιλούμε για ανάπτυξη μπορεί ο καθένα να δίνει διαφορετικό περιεχόμενο και θα ήθελα να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. σύμφωνα με εκτιμήσει των ηνωμένων εθνών αν σήμερα οι απολαυέ των εργαζομένων γυναικών σε όλον τον κόσμο αυξάνονται στο ίδιο επίπεδο με αυτών των αντρών τότε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της αμερικής θα ήταν 9% ψηλότερο της ευρωζώνης 13% και της ιαπωνίας θα εκτοξευόταν κατά 16%. Εν αυτό δεν συμβαίνει γιατί θα σήμαινε ότι κάποιοι θα έβλεπαν τα κέρδη τους να μειώνονται. Και αυτό είναι απόδειξη ότι το κυριότερο που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιο είναι το κριτήριο και το μέτρο μας. Τα κέρδη ή οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Έχουμε 11 ομιλητές στον κατάλογο ομιλητών. Θα ξεκινήσουμε με τους πέντε πρώτους βουλευτές και μετά θα απαντήσουν οι δύο επίτροποι στην πρώτη, στον πρώτο αυτό ερωτήσεων. Και μετά θα περάσουμε στους επόμενους. Ο κύριος Ντόμπρ, πρώτα απ' όλα, από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, μέλος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνική Προστασία. Και μετά ο κύριος Ζεύβιν θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντόμπρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά. Σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων, αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων. Είναι κάτι πολύ βασικό και για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τις χώρες μέλη εκεί όπου πάνε. Η κινητικότητα λοιπόν των εργαζομένων δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την ενιαία αγορά. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα άρθρο στη συνθήκη που αφιερώνεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν η Ρουμανία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς σκεφτήκαμε ότι για μας είναι πολύ σημαντικές οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλαμε να τις εφαρμόσουμε. Το θέμα λοιπόν της ελεύθερης μετακίνησης είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιπτώσεις άμεσα πάνω στον κόσμο, στους πολίτες. Η τήρηση λοιπόν αυτής της αρχής, ο σεβασμός αυτής της αρχής σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να χαίρει αξιοπιστία. Γι' αυτό λοιπόν και είναι πάρα πολύ απογοητευτικό που 10 χώρε μέλη αποφάσισαν να ε, διατηρήσουν τους περιορισμούς όσον αφορά την μετακίνηση εργαζομένων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ενώ στη συνθήκη προσχώρησης μας είχαμε δύο μεταβατικές περιόδους για τους ε, εργαζόμενους προέλευσης αυτών των δύο χωρών που θέλαν να πάνε να δουλέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εφόσον, και αν και εφόσον εκείνη η άλλη χώρα ήθελε να εφαρμόσει περιορισμούς. Όμως, για το τελευταίο στάδιο, μέχρι το 2013, αναφέρονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί η χώρα η οποία επιθυμεί να εξακολουθεί να διατηρεί περιορισμούς. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν προβλήματα στην αγορά εργασίας ή αν εντοπίζονται απειλές. Όμως, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου του 2011 δείχνει ότι η κινητικότητα δεν είχε ποτέ αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας των χωρών μελών. Καθ' άλλο, η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων είχε μόνο θετικές επιπτώσεις. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε οι δέκα αυτές χώρες να αναθεωρήσουν την στάση τους και να τηρήσουν τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητικότητα των εργαζομένων δεν πρέπει να αποτελέσει θύμα λαϊκιστικών εξάρσεων. Εμείς υποστηρίζουμε τις ε, αρχές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου που μας πέρασε το δείχνουν ε, πόσο πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφωνεί με τις αρχές αυτές και είναι κάτι που εκτιμούμε όλος ιδιαίτερως εμείς στη Ρουμανία. Τέλος, προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε δύσκολους καιρούς. Αποφασίσαμε να μοιραστούμε τις ευθύνες με τις χώρες μέλη. Εμείς θα συνεπογράψουμε τη νέα συνθήκη μαζί με τα μέλη της Ευρωζώνης αλλά πιστεύω ότι από την άλλη μεριά πρέπει να μας αντιμετωπίσετε επί ίσης ώρες. Να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ελεύθερη η μετακίνηση των εργαζόμων αποτελεί μία αξία που οι περισσότεροι βέβαια από εμά ερμηνεύουμε όπως θα έπρεπε. Ο κύριος Βιμπτόρα, Σλοβενία, είσαστε μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Κοινοβουλίου σας και μετά η κυρία Σανσές Καμασό από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ κύριε Σανίν. Ε, εγώ είμαι νέος βουλευτής και κατανοώ την αρχή αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης ως μια ατέρμονη αρχή. Ε, ανάπτυξη δηλαδή και σε καλούς ε, καιρούς και σε άσχημους μπορεί στους άσχημου καιρού να είναι μικρότερη ανάπτυξη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είναι ανάπτυξη και πρέπει να είναι φιλική προ το περιβάλλον. Η σύγκληση των ε, κρατικών ε, προπολογισμών είναι προφανώ σημαντική, έτσι ώστε να υπάρξει πάλι αξιοπιστία προ τι χώρε μα. Το θα είναι λοιπόν πιο, ε, πιο φτηνό και για του πολίτε το χρήμα και για τις τράπεζε. Μόνο που η σύγκληση αυτή πρέπει να γίνει σε πραγματικέ καταστάσει, σε πραγματικέ συνθήκε, χωρί να δημιουργηθεί μεγαλύτερο σοκ στην οικονομία. Η σύγκληση αυτή θα πρέπει να γίνει για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και να γίνει με δίκαιο τρόπο. Βεβαίω οι πιο φτωχοί θα πρέπει να εξαιρεθούν. Σε τέτοιου καιρού σύγκληση δεν μπορούμε ας πούμε, να μειώσουμε του φόρου, στην ε, Σλοβενία τουλάχιστον, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι ώστε να ενισχύσουμε τι υποδομέ ή να δημιουργήσουμε νέε. Καλό λοιπόν θα ήταν ε, αν μπορούσαμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ κατά μία μονάδα. Ε, στην ε, Σλοβενία βεβαίω ε, ο ΦΠΑ είναι, είναι σχετικά χαμηλός, οπότε αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια λύση που θα είχε βεβαίως και επιπτώσεις και στην οικονομία. Ε, βεβαίως αυτό δεν θα πλήξει τους ε, πιο φτωχούς, ε, γιατί εκεί θα υπάρξει πιο χαμηλός συντελεστής. Ε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ότι, ώστε η οικονομία να, έχει, να μπορεί να κινείται με τα, με κονδύλια που έχει. Επίσης, η ενέργεια πρέπει να παράγεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Και επίσης πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες μας ότι πρέπει να ζουν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να χρησιμοποιούν την, μια φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, θα διευκόλυναν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα βοηθούσαν την κοινωνία να πάει ένα βήμα παρακάτω. Μία λογική λοιπόν ε, σύγκληση αυτή ε, των, κρατικών οικονομικών σημαίνει πιο φτηνό χρήμα και για τις τράπεζες και για τους πολίτες και θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες μας για να κατανοήσουν και να το κάνουν εκτίματος ότι πρέπει να ζουν με πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπο. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση που κάνατε και τη συμφορά αυτών των πτυχών που θίξατε. Δεν ξέρω αν μπορεί να βάλετε ένα ΦΠΑ μεταβλητή ανάλογα με τις κατηγορίες εισοδημάτων των πολιτών. Περισσότερο κατά κατηγορία αγαθών μπορεί να γίνει αυτό. Η κυρία Σάντσε Καμάτσο τη Ισπανική Γερουσία Μέλλον τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνική Ασφάλεια Ασφάλισης και μετά και ο Ρμπιγιούν. Η κυρία Σάντσες Καμάτσο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους επιτρόπους για αυτά που είπαν. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς που ακούσαμε νωρίτερα, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εγώ είμαι από την Γερουσία της Ισπανίας και πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα που συζητάμε, που είναι η τήρηση των συνθήκων και θέμα για το οποίο πρέπει να συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργαζόμενοι και εξετάζοντας από κοινού τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές. Έχει τεράστια αξία. Όταν ε, εμείς μεταφέρουμε τις, τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα σε εθνικό επίπεδο, η πράξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό χρειάζονται τέτοιες συναντήσεις σαν τη σημερινή. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Ισπανία, όπω γνωρίζετε, υποφέρει από ιδιαίτερη υψηλή ανεργία. Έχουμε 5.300.000 ανθρώπου οι οποίοι θέλουν αλλά δεν βρίσκουν δουλειά. Τα επίπεδα επίση ανεργία στου νέου είναι τη τάξη του 40% και σε ορισμένα σημεία τη Ισπανία είναι πάνω από 54%, φτάνουν ακόμα και το 60%. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη χαμένη γενιά. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειαζόμαστε επιγόντω ε, μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ στους δύο επιτρόπους οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει το κοινωνικό ταμείο. Ο, μερικές φορές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα αυτά σε κάποιες χώρες, μήπως μπορεί να βρεθεί τρόπος ε, σε άλλους στόχους να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά. Τις τελευταίες αυτές εβδομάδες έχουμε περάσει τρεις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις διαφθορτικού χαρακτήρα. Την οικονομική μεταρρύθμιση, την εργασιακή μεταρρύθμιση και περάσαμε επίσης και μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι η εργασιακή μεταρρύθμιση ήταν ε, απόλυτα αναγκαία, ιστορική σημασία, γιατί έτσι παρακάμπτουμε μια ε, δύσκολη κατάσταση από τις πιο δύσκολες που είχαμε στις χώρες του ΟΣΑ, μια άκαμπτη κατάσταση. Σε θέματα επίσης συμβάσεων για νέους κάτω των 30 ετών ή για άτομα πάνω από 40 που δύσκολα μπορούν να επανανταχθούν στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνονται και μέτρα που έχουν να κάνουν με την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας στην Ισπανία. Εσείς λοιπόν τι βοήθεια πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εξάντε ή τι θα μπορούσαμε ε, να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Εγώ ήμουν υπεύθυνη στην προηγούμενη θητεία, στην προηγούμενη θητεία όπου κυβερνούσε το Λαϊκό Κόμμα. Μπορέσαμε τότε να ε, φτιάξουμε το Ισπανικό Θαύμα με 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι ο εθνικός προπολογισμό που πάει στις επενδύσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις περιπτώσεις αυτές που σας ανέφερα, μια που η Ισπανία χρειάζεται εκτός από τις μεταρρυθμίσεις και την άμεση αυτή βοήθεια και για μέχρι το 2020, αλλά και άλλη βοήθεια η οποία θα έπρεπε να δοθεί ευθύ αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο οριτές θα ακούσουμε, μετά θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. κύριο Μισελ Ερμπιγιόν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως μετά ο συνάδελφός μου Γκόραν Φάρμ. Ε, Κύριε Σερμπιγιόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε στην Ολομέλεια ε, στις διάφορες ε, δημοσιονομικές διαδικασίες και θεωρήσαμε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Ταυτόχρονα όλοι συμφωνούν ότι η διαδικασία αυτή του προπολογισμού δεν είναι αυτός σκοπός. Στόχος είναι η ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Έχω μία απλούστατη ερώτηση και περιμένω μία απάντηση προφανώς που να μην αντιστοιχεί, να μην εκφραστεί σε ξύλινη γλώσσα από τους συνομιλητές μας. Τι γίνεται με τη στατηγική Ευρώπη 2020, ο πρόεδρος Μπαρόσο αναφέρθηκε στο θέμα, αλλά έχουμε την εντύπωση και ίσως ε, θα τα απορρίψετε αυτό, ότι λόγω της κρίσης του ευρώ, λόγω της ελληνικής κρίσης, λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, λόγω των διαπραγματεύσεων της νέας συνθήκης, εν συντομία λόγω της οικονομικής κρίσης, η στρατηγική Ευρώπη του 2020 ενδεχομένως έχει μείνει στο περιθώριο για να μην πούμε ότι ανεβλήθη, μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας πέρα το 2020. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ελπίζω προφανώς να μην είναι κάτι τέτοιο που ισχύει, θα ήθελα να μας πείτε ενδεχομένως οι επίτροποι να μας πούν πώς μεταφράζεται αυτή η στρατηγική Ευρώπη 2020 σε συγκεκριμένες ευανάγνωστες πράξεις με έναν τρόπο αντιληπτό για τους πολίτες μας, συμπολίτες μας. Ήτι οι συμπολίτε μα στι διάφορε χώρε Ευρώπη να μπορούν να εστερνιστούν αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική. Είδεμη, φοβούμε ότι, ότι ε, το πρόγραμμα Ευρώπη του 2020 μήπως μοιάζει πολύ με στρατηγική της Αβώνας που τελικά και το λέω μεταθλίψεως αυτό ε, ήταν ένα συνεχές ευχολόγιο που δεν μεταφράστηκε σε πράξεις και σε συγκεκριμένα μέτρα για τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τελευταία ομιλία όσον αφορά την πρώτη αυτή παρτίδα. Ο κ. Γκόραν Φάρμ, ένας από τους τέσσερις συγητές της Επιτροπής Προπολογισμών για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, είναι ευρωβουλευτής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ναι, ναι. Και είμαι και συγητής του Κοινοβουλίου για τα project bonds, για την πιλωτική φάση αυτών των ομολόγων. Αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να αφαιρθώ σε μία ομιλία Σουηδού συναδέλφου του Σουηδικού Κοινοβουλίου στο Ενολομέλεια. Είναι συντηρητική και είπε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε επί της λιτότητας και να μην, ε, να, παρετηθ, να μην ανταποκριθούμε σε κλήσει για τον της οικονομίας και να επανέλθουμε γρήγορα στην σωροπία. Δεν συμφωνώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Σουηδία ως ένα παράδειγμα του γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα. Είχαμε μεγάλη κρίση αρχή της δεκαετίας του 90 Σουηδία, κατέρευσαν τράπεζες κλπ καταφέραμε να βγούμε μέσω πολύ περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων και όχι μόνο αυτό, καταφέραμε να διατηρήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του συστήματος του δημοσίου και το σύστημα πρόνοιας. Κάναμε τις μεταρρυθμίσεις, τα διατηρήσαμε αυτά. Διατηρήσαμε φιλόδοξους στόχους παιδείας ε, και αγοράς εργασίας για να αποφύγουμε το υψηλό επίπεδο ενεργείας. Αποφασίσαμε επί μακροπροθέσμων στρατηγικών για να επανέλθουμε στην ισορροπία και χρειαστήκαμε από μείον 11% για να πάμε από ένα έλλειμμα 11% του ΑΕΠ να το εξορροπήσουμε χρειαστήκαμε 7-8 χρόνια και όχι ένα ή δύο και κάναμε και κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα διότι ζητήσαμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε ε, και αυτό βοήθησε πολύ. Τι θέλω να πω, χρειαζόμαστε ισορροπημένη στρατηγική όχι μέγιστη βραχυπρόθεσμη λιτότητα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε μια κατάσταση όπω αυτή που επικρατεί στην Ελλάδα σε ένα-δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε συνεργασία στην Ευρώπη, επενδύσει σε μια πραγματική έννοια αγορά, να χρησιμοποιήσουμε το ότι είμαστε 500 εκατομμύρια καταναλωτέ, Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Αυτοί που είναι σε καλύτερη θέση θα πρέπει να είναι έτοιμοι να επενδύσουν για να βοηθήσουν και του εαυτού του και του άλλου. Και γι' αυτό η περικοπή του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι λύση. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τώρα που θέλουν να περικόψουν 100 δι από τι επόμενε δημοσιονομικέ πολιτικέ, περίπου 10%. Διότι αν το κάνουμε αυτό, μόνο τα κράτη που είναι καθαροί συνεισφορεί θα ωφεληθούν. Ενώ εκείνοι που χρειάζονται τα χρήματα θα χάσουν. Το ερώτημά μου απευθύνεται και προ εθνικού βουλευτέ και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ πείθουμε τα κράτη που συνεισφέρουν στον προπολογισμό, τα προγράμματα, τα εθνικά ταμεία, τα project bonds, όλα αυτά οι επενδύσει είναι χρήσιμα και για του συνεισφορεί και για του αποδέκτε. Διότι αν δεν μπορούμε να του πείσουμε, φοβούμε ότι η διαδικασία του προπολογισμού ή τη επόμενη δημοσιονομική προοπτική θα προσθέσει στη λιτότητα παρά το αντίθετο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να ακολουθήσετε την ίδια σειρά στις απαντήσεις ο Επίτροπος ο κ. Λεβαντόφσκι, πρώτος ίσως. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και θα ξεκινήσω από τον κύριο Ντόμπερτς από τη Ρουμανία. Η κινητικότητα είναι ένα κομμάτι της ελευθερίας της ενιαίας αγοράς. Τώρα στη σκιά της κρίσης βέβαια βρίσκεται. Είναι στόχος θεμητός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ξέρω ότι υπήρχαν περιορισμοί που αντικατόπτριζαν και κάποιες προκαταλήψεις περί εισβολής των δυτικών αγορών εργασίας από εκείνους που βρισκόταν πίσω του σιδηρούν παραπέτας. Ίσως είναι θεμητή η φόβη σαν απάντηση στις ανησυχίες του πληθυσμού της Δυτικής Ευρώπης. Βεβαίως όμως αυτές οι απόψεις είναι αντίθετες προς μία από τις καθαγιασμένες ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όσον αφορά την κινητικότητα, δοθήσεις της εμπειρίας άλλων χωρών, όχι της Ρουμανίας, η κινητικότητα θα μπορούσε να είναι και μονόδρομος. Θα μπορούσε να είναι μονόδρομος. Που ανθρώπους που αρπάζουν τις ευκαιρίες εκεί που υπάρχουν καλύτερες πληρωμές και δεν επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Δύο φορές τουλάχιστον Πήγα σε δύο νέα κράτη-μέλη. Και ζητήθηκε εκεί να μην προωθείται πολύ το πρόγραμμα κινητικότητα ή την νεολαία, διότι ήδη κινείται η νεολαία, ξεφεύγει. Μου να μην το, ζήτησα να μην το προωθούμε, να μην ξεγλιστράει, να μην ξεφεύγει η νεολαία, διότι δυστυχώ ε, αυτή η μετακίνηση είναι μονόδρομος, λόγω των διαφορών των αμοιβών. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιμείνει επί της πλήρους εφαρμογής ε, τη σημαντική αυτής ελευθερίας, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, όμως έχω σωρεύσει μεγάλη εμπειρία σε διάφορα κράτη-μέλη, βλέποντας ότι αυτό δεν είναι τόσο καλό και δεν είναι υποφελή κατάσταση για όλους. Είναι ένας μονόδρομος περισσότερο και δεν είναι μόνο μια προσωρινή κινητικότητα. Όσον αφορά το ερώτημα της Σλοβενίας ε, για τη φορολόγηση. Τι γίνεται στα διάφορα θεσμικά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο να κάνουμε πρόταση. Βάση, δεν υπάρχει, βάση το ότι δεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση άνευ εκπροσώπηση. Και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την αρχή. Ακόμα και αν προτείνουμε άλλες πηγές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για πόρους, ε, τελικός λόγος ανήκει στα εθνικά κοινοβούλια είναι προνόμιο ομόφωνης απόφασης των κρατών μελών, κύρωση στα κρατη ε, στα κοινοβούλια, συγγνώμη, και εγώ θα κάνω πρότηση για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και στα πλαίσια και του ΦΠΑ σαν ένα κομμάτι των εισόδων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είναι μέτρο που θα πρέπει να επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρία Σάντσες Καμάτσο. Γνωρίζω καλά την κατάσταση που κρατεί τώρα στην Ισπανία. Την περασμένη εβδομάδα μια ειδική ομάδα πήγε στην Ισπανία για να συζητήσει με την κυβέρνησή σας και τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη πώς να γίνει ένας αναπρογραμματισμός των διεθνωτικών ταμείων προς όφελος των θέσεων απασχόληση να δημιουργήσουμε θέσεις για τους νέους. Ο Χάν καταφθάνει στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα για να το συζητήσει το θέμα. Τώρα έχει ανάψει πράσινο φως. Υπάρχει μια δυνατότητα αναπρογραμματισμού για να δημιουργηθούν δυνατότητες απασχόλησης σε χώρες όπως η Ισπανία. χάνει κάποια, κάποιοι τομεί χάνουν την επιλεξιμότητα για στήριξη από τα περιφερειακά ταμεία, αλλά είναι περιοχή σύγκληση ακόμα η Στρεμαδούρα. Η Μούρθια, η Γαλήσια, η Λαμάντσα και άλλε. Η Ανδαλουσία πάνω απ' όλα. Είναι ενδιάμεσες περιοχές ε, με αρκετά εντατική βοήθεια που δέχονται. Ε, οπότε αντίθετα με τα στερεότυπα που ακούγονται στην Ισπανία ότι θα συνεισφέρει, θα είναι ξεκάθαρα συνεισφορέ τη Ισπανία στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αντιθέτω, ε, θα εξακολουθεί να είναι δικαιούχο βασικό και να ωφελείται από τα προγράμματα Ισπανία. Τρευλό τρόπο να μετρήσει κανεί την επιτυχία όταν από δικαιούχο μια χώρα αποδέκτη γίνεται συνεισφορέα. Το κοινωνικά ταμεία απορροφήθηκαν σωστά από την Ισπανία πέρσι. Η 111% απορρόφηση είχαμε στην Ισπανία από αυτά που προβλεπόταν για το 2011. Και όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν την αγορά εργασίας στην Ισπανία. Σύμφωνα με τη σειρά που έθεσε η κυρία Πρόεδρε, στα δύσκολα ερωτήματα θα τα απαντήσει ο Ιωάννης Χάν. <laughs> Ε, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον ε, ε, Ευρωβουλευτή Φάρμ για την παρουσίασή του. Είπε ο ίδιος ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ε, θα συμφωνήσω με αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πρέπει όμως να εργαστούμε σκληρά ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση αλλά θα ήταν άδικο να πούμε ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μέσα σε λίγους μήνες ε, θα μπορέσουμε την ανεργία των νέων να την αντιμετωπίσουμε βιώσιμα, ή να τη μειώσουμε βιώσιμα. Ε, μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα μπορούμε να κάνουμε αρκετά, αλλά το θέμα είναι αν είναι παρκώς βιώσιμα όλα αυτά που κάνουμε. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να δρούμε με έξυπνο τρόπο και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας βιώσιμες και για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενισχύσουν και αυτές την δυνατότητα καινοτομία που έχουν. Βεβαίως και στο θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να ενισχύσουμε τον τομέα αυτό. Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία και η επαγγελματική κατάρτιση Συνήθως ε, ε, στην επαγγελματική κατάρτιση υπάρχει ε, ανισορροπία μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής γνώσης. Οπότε πρέπει να δούμε αν οι θεωρητικές γνώσεις που προσφέρονται τελικά απαντούν και στις ανάγκες της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο, μεγα, πιο αυξημένες ταχύτητες απάντησης, ανταπόκρισης. Για παράδειγμα όμως θα μπορούσα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη έχουμε 23 ε, εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε και 23 εκατομμύρια ανέργους. Αν λοιπόν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούσαν να προσλάβουν έναν ακόμα εργαζόμενο θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Αν τώρα το αφήσουμε ε, στο, στις 500 ε, ε, μεγαλύτερες επιχειρήσεις να προσλάβουν υπαλλήλους, θα έπρεπε ο κάθε μία από αυτές τις 500 μεγάλες επιχειρήσεις να προσλάβουν 46.000 ανθρώπους για να λύσουμε το θέμα των 23 εκατομμυρίων ανέργων. Οπότε προφανώς είναι πιο απλό να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι γίνεται και με την εξειδίκευση, την έξυπνη εξειδίκευση πρέπει και σε αυτό το τομέα να δούμε ποιε είναι οι υποδομέ που υπάρχουν και να τις ε, αναπτύξουμε με έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και αγορές εργασία, οι οποίες θα είναι βιώσιμες. Ε, εμένα είναι από κοινού με τα κρατημέλη να δημιουργήσουμε δυνατότητες και εν τω μεταξύ θα μπορούσα να σας πω, ε, μια που έχω επισκεφθεί ήδη πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη, ότι παντού σε κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη υπάρχει μία ειδικότητα σε μια, ή μια εξειδίκευση σε μια περιφέρεια την οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε έτσι ώστε να, γίνουν, να δημιουργηθούν βιώσιμες ε, θέσεις εργασίας. Τώρα για την Ευρώπη 2020 δεν έχει πεθάνει, το αντίθετο είναι ζωντανή και πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Και εδώ πάλι έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πόσο απαραίτητη είναι ε, αυτή η, πόσο απαραίτητο είναι ο πολυετής προγραμματισμό σε οικονομικό επίπεδο για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και να θέτουμε σωστού στόχου. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι συγγνώμη, στο πώ θέτουμε του ε, στόχου μα. Θέλουμε όμω να μειώσουμε την ε, ανεργία. Αυτό είναι ένα στόχο. Θέλουμε να μειώσουμε τα παιδιά που φεύγουν από τα σχολεία πριν ολοκληρώσουν την, ε, την ε, εκπαίδευσή τους χωρίς πτυχίο. Ε, αυτό προφανώς πρέπει να αποτελεί στόχο μας. Θέλουμε να αυξήσουμε τους εξειδικευμένους επιστήμονες, θέλουμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε τελικά τις, ανεργία, τις ανανεώσιμες ενεργείες να τις ενισχύσουμε. Αυτά είναι κεντρικοί στόχοι, οι οποίοι παραμένουν. Είναι αδιαπραγμάτευτοι στόχοι και πρέπει να ενισχυθούν μέσω της Ευρώπης 2020. Είναι στόχοι του Ευρώπη 2020 και πρέπει να, να παρακολουθηθούν και να προωθηθούν και από το Ταμείο Συνοχής. Αυτή λοιπόν η πολιτική θα πρέπει να γίνει σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, γιατί έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια των μέτρων και να εξασφαλίσουμε επίσης ότι οι στόχοι αυτοί θα εκπληρωθούν. Και σε σχέση με αυτό και αυτό βεβαίω πρέπει να είναι ειδοποιώ διαφορά με τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Είναι απαραίτητο να είναι ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι και σε εθνικό και αν γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο. Να είναι δηλαδή φιλόδοξοι αλλά να είναι και ρεαλιστικοί. Αυτό πρέπει να το δούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες. Αυτοί οι στόχοι όμως θα πρέπει να δημοσιευθούν, να προωθηθούν προς τα έξω έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε κιόλας. για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουν τελικά συμφωνηθεί. Πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα να προχωρήσουν πιο γρήγορα, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, γιατί εδώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε προοπτική για τους νέους. Απ' την άλλη όμως πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε ειλικρινεί. Δεν μπορούμε εν μία νυχτή να περιμένουμε ότι τα προβλήματα θα λυθούν. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς προοπτικές. Να ξεκινήσουμε με την εργασία σήμερα, όχι αύριο, και ειδικά τους νέους, αλλά όλους μας τους πολίτες, να τους ε, δώσουμε ε, μια αίσθηση εμπιστοσύνη ότι το κράτος είναι εκεί και υπάρχει για να, για να λύνει προβλήματα και όχι για να δημιουργεί προβλήματα. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Μίλτ πρώτα απ' όλα από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, Είσαστε αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρει η Κρυζανίν Κάνα. Κύριε Μίλα, έχετε εσείς το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από την Ουγγαρία από την χώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το μαστίγιο, όπως είπε ο κ. Λεβαντόσκι πιο πριν. Μιλούμε για την ε, οικονομική κρίση, για τους ε, προϋπολογισμούς, ε, μιλούμε για τη σύγκληση μεταξύ των διαδικασιών, της πραγματικής οικονομίας, των ε, δημοσιονομικών στοιχείων. Μια ανάλυση αυτών των, ε, αυτής της προβληματικής θα μας βοηθούσε πραγματικά. Υπάρχουν όμως και κάποια βασικά προβλήματα. Η προσπάθεια να ρυθμιστούν ή να φορολογηθούν, να υπάρξει μαροφορολόγηση, ναι, είναι καλή, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Και μάλιστα η περιφέρεια έχει τεράστιες διαφορές σε σχέση με τις, ε, με τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση με την παραγωγικότητα, με την ανεργία κτλ. Βασικό λοιπόν ε, είναι να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε που υπάρχει, να μην ε, δημιουργούμε επιπλέον οξύνσεις. Εάν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας και της, ε, ε, των άνισων ευκαιριών που υπάρχουν για την ε, περιφέρεια, δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία Ευρώπη. Πολύ σωστά είπαν η Επιτροπή ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη φυσικά οι περιφέρειες, γιατί έχουν ειδικέ εξειδικεύσει, ειδικά, ειδικά χαρακτηριστικά, ειδικά για τις χώρες που, δεν που είναι σε πιο αδύναμη θέση, δεν απορροφούν τα κονδύλια και πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφ φως δυνατό. Και πρέπει να εμπλακούν οι χώρες αυτές. Τώρα, αν ε, μειωθούν μέσω των ε, κυρώσεων οι δυνατότητες αυτών των, ή οι πιθανότητες που έχουν αυτές οι χώρες, προφανώς μειώνουμε και, την, ε, και, το μέλλον τους και τις προοπτικές που έχουν. Δεν μπορούμε να, να τιμωρούμε ακόμη περισσότερο αυτές τις ε, χώρες. οι, βεβαίως οι χώρες που προσφέρουν τα χρήματα είναι αυτές που χάνουν και τμήμα της αγοράς. Έχουμε και κάποιες ανησυχίες βεβαίως, τις οι οποίες ήδη αναφέρθηκαν ακροφηγώ, ότι δηλαδή αυτό το, αυτή η συμφωνία δεν έγινε με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι προχωρούμε με μη δημοκρατικά μέσα. Επίσης μια άλλη ανησυχία μας είναι το σε ποιο βαθμό μέσω μόνο κυρώσεων μπορεί να υπάρξει πρόοδος, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην αγορά εργασίας. Μιλούμε για ένα σύμφωνο το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με τα βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά λείπουν πολλά στοιχεία από αυτό το σύμφωνο. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα ταμεία συνοχής, στην Ουγγαρία μιλούμε για 142 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα ήθελα να μιλήσω για ένα μόνο στοιχείο. Αν ε, το θέμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας ε, και δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις, τότε πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει, α, ε, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή που να λένε ότι η χώρα μας είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να πάυσουν αυτές οι Δεν υπάρχουν ούτε αναλύσεις, ούτε υπολογισμοί, ούτε τέτοια στοιχεία. Προφανώ ο προπολογισμό μα βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι ακραίε πολιτικές δυνάμει ενισχύονται. Ε, και κάτι άλλο για την ε, πολιτική απασχόληση στην Ουγγαρία. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, περιορίζοντας τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων και χειροτερεύοντας τις ε, σχέσεις εργασίας τους, ε, προφανώ δεν θα καταλήξουμε σε μια Ευρώπη που να είναι βιώσιμη. Πρέπει να έχουμε υποδείγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε απλώ μια διαχείριση κρίση. Ναι. Ευχαριστούμε κύριο Χάνιγκαν. Ιρλανδία. Βουλή των Αντιπροσώπων. Είσαστε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Και στη συνέχεια ο κύριος Κύριε Χάνινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε πολύ που μας δίνετε ευκαιρία να συμμετέχουμε στη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Πολλοί γνωρίζουν ότι χωρίς ε, να εξεταστεί αν χρειάζεται δημοψήφισμα ή όχι, η συζήτηση παρόλα αυτά στην Ιρλανδία έχει ξεκινήσει. Και εγώ είμαι κατά. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι για λιτότητα και μόνο για λιτότητα, χωρίς να κάνει τίποτα η Ευρώπη για την απασχόληση. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα μιλάμε για την Ευρώπη του 2020 και χαίρομαι που μιλάμε κυρίως για την ανεργία των νέων. Όπως και οι Ισπανοί, έτσι και εμείς υποφέρουμε πολύ από την ανεργία αυτή. 30% περίπου των νέων μα είναι στην ανεργία. Κάτι το οποίο όπως και στην Ισπανία και εδώ οδηγεί σε μια χαμένη γενιά νέων και σε μεγάλη μετανάστευση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στο Δουβλίνο μια ομάδα από την Ευρώπη που ασχολείται με την απασχόληση. Η ερώτησή μου είναι τα μέτρα πού θα βασιστούν. Ορισμένες ε, χώρες δεν έχουν ε, χρησιμοποιήσει ε, καλά ίσως τα διευθυντικά ταμεία, τέλος πάντων τα έχουν ξοδέψει όλα. Θέλω λοιπόν να ξέρω χρήματα από χώρες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ε, όλα τα χρήματα που πήραν για τα ορθωτικά ταμεία θα μπορέσουν να τα δώσουν ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις χώρες εκείνες οι οποίες πραγματικά τα χρειάζονται τώρα για βιώσιμη απασχόληση. Είναι ζωτική σημασία. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αν συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η δικιά μας η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα ε, πρότεινε 270 διαφορετικά μέτρα έτσι ώστε να βοηθήσει τις μικρές ε, επιχειρήσεις, να δει πώς θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, τα startups. Χρειαζόμαστε όμως και ένα σχέδιο απασχόλησης από τη δικιά σας την πλευρά, το οποίο να συμπληρώνει αυτά τα οποία κάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις και να μην τα αντικαθιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριο Σαρτούι τώρα από την Γαλλική Γερουσία παρακαλώ και μετά ο κύριος Κλαπισό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος ναι. Ερπουή από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι προσπαθούμε να έχουμε ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αλλά όλα δεν διακανονίζονται με τον προπολογισμό, χρειάζονται και διορθωτικέ μεταρρυθμίσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να συντονίσουμε τις ε, πρωτοβουλίες και να συναντηθούμε κάπου έτσι ώστε να συνεργαστούμε πάνω σε διάφορες δράσεις. Όσον αφορά τον προπολογισμό, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις, παρακαλώ. Πρώτον, στα δημοσιονομικά θέματα, το βασικό των δημοσίων δαπανών το αναλαμβάνουν οι χώρε, Οι χώρε το αποφασίζουν δηλαδή και ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό, όσο μεγάλο και αν είναι, είναι τελικά περιθωριακό. Πρόκειται για 2% περίπου των δημοσίων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, καλό είναι να αντιληφθούμε καλύτερα την πραγματικότητα των δημοσίων δαπανών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα ήθελα να τυποποιήσουμε τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε και τις μεθόδους με τις οποίες παρουσιάζουμε τα δημοσιονομικά των χωρών για να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια. Τι να τους κάνουμε τους χρυσούς κανόνες αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Και τέλος πρέπει τους λογαριασμούς μας να τους παρουσιάζουμε σε δισεκατομμύρια ευρώ και όχι βάση του ΑΕΠ. Γιατί αν θέλουμε να δούμε ολόκληρο τον προπολογισμό αυτό πρέπει να κάνουμε. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει επαρκή συντονισμός, ότι υπάρχει μεγάλη ανισορροπία και ότι άρα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα και να συνεργαστούμε καλύτερα πάνω στις εθνικές μας πρωτοβουλίες και να τις συντονίσουμε με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση των χωρών εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σε αντίθεση με τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλλά δεν είναι στην Ευρωζώνη, στην Ευρωζώνη τα πράγματα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Άρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ιδιαίτερο τρόπο τα διευθυντικά ταμεία. Γιατί αν δεν γίνει αυτή η προσαρμογή και αν ψάχνουμε αυτοχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο, παραπάνω έλλειμμα ε, θα έχουμε τη στιγμή που ήδη υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και χρέωση. Και να εκφράσω και μια ευχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι υπάρχει μια στρέβλωση και μια αντίφαση ανάμεσα στις ανησυχίες της εσωτερικής αγοράς και τις ανησυχίες της Ευρωζώνης. Η εσωτερική αγορά ε, φτιάχνει κανονισμούς, οδηγίες που επιταχύνουν τις δημόσιες δαπάνες ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Ενώ μέσα στην Ευρωζώνη θέλουμε την οικονομική σταθερότητα, την μείωση των ελλημάτων, της χρέωσης, την εξυγίανση των δημοσιονομικών και περισσότερη ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν και αυτή είναι η ευχή μου να εναρμονίσουμε κάποια στιγμή τις ανησυχίες αυτές και να συμφιλιώσουμε μέσα στην εσωτερική αγορά τους παραγωγούς με τους καταναλωτές. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κλαπισού της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, απειχώντας τα όσο είπε ο Αχτουή, να υπενθυμίσω την παράγραφο 33 του πρόσφατου κειμένου επί του θέματος που ψηφίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκαν πολλά κείμενα σχετικά, διότι είναι μόνιμη ανησυχία και των Ευρωβουλευτών αυτή. Στην έκθεση του κ. Γκοζέ, παράγραφο 33, καλείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να επεξεργαστεί πραγματική κοινή ονοματολογία όσον αφορά τα λογιστικά και τον προπολογισμό, ούτω ώστε όλα αυτά να γίνεται συμπλήρωση, πρόσθεση των ε, εξόδων για να μπορεί να χρησιμοποιείται εθνικό προπολογισμό και ευρωπαϊκό προπολογισμό για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων. Ο κύριο Κάπισον της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μετά η κυρία Ζαχτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή την συνάντηση. Είναι μεγάλη ευκαιρία να ανταλλάσσουμε εμείς απόψεις οι εθνικοί βουλευτέ και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Και ίσω να διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ με κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό να γίνονται αλλαγή απόψεων, ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε την κατανόησή μα όσον αφορά τι πεπιθήσει μα. Όσον αφορά το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, αυτό δεν είναι το βασικό σημείο. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι το μέγεθο του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι τέτοιο που δεν θα ήταν ρεαλιστικό να δούμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που θα μπορεί να αντισταθμίσει μακρο, μακροοικονομικά προβλήματα. Και υπάρχει κάτι άλλο και προσέξτε το, ε, κύριε Σουηδέ, συνάδελφε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κανεί αυξήσει για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και για τη δίκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για τα προγράμματα δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνουν πάρα πολύ σημαντικέ ε, ε, περικοπές στα δημοσιονομικά τους. Ζητάμε από τον κόσμο να δεχτεί μείωση των δαπανών, που αυτό έχει συνέπεια στην απασχόληση, μείωση υπηρεσιών, κυρίως σε κάποιους τομείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει δημοκρατική συμφωνία για αύξηση δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη από αυτό. Το βασικό που θέλω να πω όμως δεν ήταν αυτό, είναι κάτι άλλο. Αφορά το μέλλον του ευρώ και την πολιτική που περιγράφτηκε σήμερα και η οποία υπονοείται στο νέο σύμφωνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο ευρώ προφανώς, αλλά εξίσου προφανώς θέλουμε να δούμε σταθερότητα στην Ευρωζώνη και θέλουμε να δούμε ανάπτυξη και ευημερία στον ευρωπαϊκό χώρο. Ακούσαμε σήμερα το δρομολόγιο που προτείνεται, την πορεία που προτάθηκε. Απευθύνω έκκληση προς εσάς. Δείτε αυτή την προσέγγιση να είστε σίγουροι ότι λειτουργεί. Και αν δεν λειτουργεί, ας είστε ανοιχτοί να αλλάξετε πορεία. Και πρέπει να πω ότι η αξιοπιστία των όσων προτείνονται δεν είναι μεγάλη, δοθέντος του υποβάθρου. Θυμόμαστε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, τα κριτήρια του Μάστρικ και τα διάφορα κριτήρια που είχαν καταρτιστεί τότε, πώ παραβιάστηκαν το παρόν σύμφωνο έχει διαφορετικές διατάξεις, διαφορετικές προδιαγραφές που περιέχει, αλλά ποιοτικά είναι το ίδιο από πολλέ πλευρές και διερωτώμεθα κατά πόσο αυτό θα επιφέρει την επιτυχία που δεν επέφερε το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη. Ακούσαμε επίσης κάτι πολύ παλιό, ε, προτάσεις για ανάπτυξη ε, που θα τονώνται από σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα τη Αβώνα και όλα αυτά. Αν τα πιστεύαμε αυτά τότε, ε, δεν θα είχαμε τα προβλήματα. Αν ισχύαν αυτά και λειτουργούσαν, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε ανάψει και την απασχόληση σήμερα. Η πολιτική προτείνεται πριν να είστε σίγουροι ότι λειτουργεί. Εγώ ανησυχώ ότι γίνεται με τα μέτρα λιτότητα που φαίνεται ότι επιβάλλονται στι χώρε τη Νότια Ευρώπη, διότι πρέπει να ανταγωνιστούν με ισοτιμίε που δεν είναι ανταγωνιστικέ για αυτού και δεν ελέγχουν οι χώρε αυτέ τα δικά του επιτόκια. Δοθέντω ότι βλέπουμε τεράστιε αυξήσει όσον αφορά την ενεργεία, πολύ ψηλά επίπεδα ενεργεία ε, στου νέου, όπω ακούμε στην Ισπανία, συνάδελφο, μείωση 7% το χρόνο στο ελληνικό ΑΕΠ. Αν έχουμε λιτότητα και θέλουμε δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα και μόνο, βλέπουμε τι συμβαίνει στι νότιε χώρε τη Ευρώπη. Θα καταρρεύσουν τα φορολογικά του έσοδα, διότι πολύ λίγοι θα εργάζονται, αύξηση των θα πάνε στην κοινωνική ασφάλιση, θα έχουν τεράστιε κοινωνικέ εντάσει και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγματι αυτέ οι χώρε να επανέλθουν σε οδήποτε ισορροπία, εξισορροπημένο, συλλογισμένο προπολογισμό. Και το λέω συντηρητικό που πιστεύει εν γέννη στη δημοσιονομική πειθαρχία σε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο. Και όσο πιο πολύ τα ακούω όλα αυτά, τόσο πιο πολύ πιστεύω ότι δεν μάθαμε κάποια τα μαθήματα τη δεκαετία του 30 όταν ακολουθήθηκαν σε κάποιε χώρε τον ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Δυτική Ευρώπη, αρχέ τη δεκαετία του 30 αυτά τα μέτρα, χωρί να έχουν φανερέ επιτυχίε μέχρι ότου που ακούσαμε από τον Κέιν διαφορετική άποψη. Λοιπόν, να είστε έτοιμοι να ξανασκεφτείτε το θέμα και θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Διακόπτη πρόεδρο. ευχαριστεί τον ομιλητή. Η κυρία Σαχτιέ και μετά κλείνω το λόγο των ε, ομιλητών και θα ακολουθήσει ένας τελευταίος γύρος πέντε μελών. Η κυρία Ζαχτιέ που είναι η εισηγήτης αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, στην, ε, σύμφωνα με αυτά που μόλις παρουσιάστηκαν, από τον συνάδελφο Ζαν Αχτουί όσον αφορά τη δημοσιονομική σύγκληση που απαιτείται με μια κοινή ονοματολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήθελα να επιμείνω επί της ανάγκης που υπάρχει να συγκλίνουν κατά πολύ οι πολιτικές απασχόλησης. Όμως αυτές οι πολιτικές είναι πολιτικές ουσιαστικά ε, εθνικής ευθύνης. Και βλέπουμε ότι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και πάνω απ' όλα να προετοιμάσουμε όλους τους μισθωτούς για την αλλαγή των προσόντων που απαιτούνται, την αλλαγή των θέσεων εργασίας, κάτι που θα χρειαστεί στο μέλλον. Ε, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε απλώς όσον αφορά την αρχική κατάρτιση, αλλά επίσης μαζί με τους μισθωτούς, μαζί με τους εργαζόμενους, όλους τους συμμετέχοντες, μαζί με τους επαγγελματικούς κλάδους θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις ζωντανές μας δυνάμεις για να προετοιμάσουμε τους εργαζομένους για τις νέες ανάγκες ε, των επιχειρήσεων. Δεν είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρόλο που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης που θα μπορέσουν να το πετύχουν μόνες τους αυτό, άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξουν τη βούληση αυτή που υπάρχει στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως μέσω των εργαλείων που υπάρχουν από τα κοινωνικά ταμεία. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν που θα πρέπει να μας εγκαταλείψει και μετά στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι που θα μείνει μαζί μας και θα απαντήσει. Πριν δώσω όμω το λόγο στον Επίτροπο Χάν, θα ήθελα εκ νέου να καταχραστώ τη θέσεις του Προέδρου Και να πω το εξή, μα είπατε αρχικά ότι στις χώρες όπου το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το πιο χρήσιμο, ε, δεν καταναλώνται, δεν απορροφούνται οι πόροι αρκετά. Ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε να διευκολυνθεί η κατανάλωση, έχουμε τον κοινωνικό διάλογο, έχουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, έχουμε μηχανισμούς μόνιμης κατάρτισης είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ίσως για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο βέλτιστο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και ίσως στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει αυτές τις δυσκολίες να τις λάβουμε υπόψη. Σαν στοιχείο του προγραμματισμού θα πρέπει να λάβει η χώρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο, διότι δεν είναι στις ε, αρμοδιότητές μου τις βασικές. Αναφέρθηκα στα στατιστικά στοιχεία, θα αναφερθώ στα στατιστικά στοιχεία με τα οποία ασχολούμαι. Αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός όσον αφορά το μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται είναι αμεληταίο ποσό. Αυτό δεν αληθεύει όμως, διότι σε πολλές χώρες τα διαθετικά ταμεία, πιο συγκεκριμένα αποτελούν σημαντικό τμήμα των δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε χώρες όπου πάνω από το 50% των δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιείται ε, μέσω των διευθυντικών ταμείων. Ακόμα και στη Γαλλία. Τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας πάνω από 50% του δυναμικού επενδύσεων στις περιφέρειες αυτές προέρχεται από θετικά ταμεία. Λοιπόν, σε πολλές περιοχές, πολλές περιφέρειες χορηγούνται διαστοτικοί πόροι, λειτουργούν καλά οι περιφέρειε και αυτέ που λειτουργούν καλά οι περιφέρειε χρησιμοποιούν τα διαστοτικά ταμεία. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε η παροχή των πόρων αυτών, διότι είναι από τους καλύτερους τρόπους για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων και για την υλοποίηση νέων ιδεών. Διότι πολύ συχνά ο δικός τους προπολογισμό, οι δικοί τους δημόσιοι πόροι είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και είναι, έχουν δεμένα τα χέρια όσον αφορά την χρήση των πόρων και τα δικά ταμεία είναι το μόνο που τους απομένει. Και βέβαια χρειάζεται να προσφέρουμε εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις που άνε ούτως ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε ιδέες σε όλη την Ευρώπη και να είμαστε συνεπείς στην προσέγγιση. Και σας λέω ανοιχτά ότι την ανάπτυξη σε διάφορους τομείς δεν θα μπορέσουμε να την κινητοποιήσουμε χωρίς χρήματα. Αν ας πούμε μπορώ να προτείνω στους, Έλληνες, στους Έλληνες συναδέλφους να σκεφτούν ότι σε κάποιες περιφέρειές τους είναι δυνατόν να υπάρξει τουρισμός όλα τα χρόνια, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ίσως αυτό, θα, αν το ασημεριστούν οι Έλληνες ε, συνάδελφοι, να μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο. Γιατί εκεί θα μπορούσαν να γίνουν ε, επενδύσεις. Ας πούμε στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων υπάρχει ανάγκη να, υπάρξει, να υπάρξουν τέτοιες δυνατότητες. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες, αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί μόνο αν υπάρξει σχετική χρηματοδότηση. Χωρίς λοιπόν οικονομικό αντιστάθμισμα αυτή η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν θα έρθει. Και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι Πώ θα γίνει, πώ θα υπάρξει αυτή η ανάπτυξη και πώς μπορέσουμε να την κινητοποιήσουμε με έναν έξυπνο τρόπο. Ε, το είπε και ο Γιάννους πιο πριν. 95% ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού πάει στα κράτη-μέλη για δραστηριότητες, επενδύεται 5%, ίσως και λιγότερο από 5% του ευρωπαϊκού προπολογισμού υπάρχει για να καλύψει τα έξοδα, τις δαπάνες, των, ε, ε τις διαχειριστικές και διοικητικές. Οπότε πρέπει να ξέρετε ποιο είναι ο λόγος μεταξύ επιχειρησιακού ε, προπολογισμού και προϋπολογισμού για τι δαπάνε. Επίσης για, τους, για το πώς καλύπτονται ή εποφελούνται οι χώρες που καταβάλουν ε, τα κονδύλια, το είπαμε και πιο πριν. Προφανώς αυτές οι χώρες εποφελούνται αρκετά, αλλά ας πούμε η Γερμανία για κάθε ευρώ που δίνει στα, στην Πολωνία μέσω των διαφορετικών ταμείων παίρνει πίσω 85 cents, 85 λεπτά για, ε, που έρχονται πίσω στις ε, γερμανικές ε, επιχειρήσεις. Απευθείας εισρωή από 1 ευρώ 85 λεπτά έρχονται πίσω στη Γερμανία. Δείχνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα για αυτό το μέσο και βιωσιμότητα, κυρίως για τις χώρες που καταβάλουν τα κονδύλια, που πληρώνουν. Για τους Ιρλανδούς συναδέλφους. Έχετε δίκιο. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε κάτι επιπλέον. Ε, ο στόχος μας είναι τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τα ανάλογα ε, προγράμματα για την ένταξη των νέων, για την αντιμετώπιση της ενεργείας τους. Ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίε ήταν και επιτυχεί. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε ίσω να το μελετήσει κάθε χώρα, να δει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή τι θεωρεί η ίδια χώρα ότι είναι ενδιαφέρον και θα μπορούσε να ε, προσελκύσει του δικού τη ε, νέου. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ε, ε, ε, χρήματα που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο στο τέλος της προγραμματικής περίοδου μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν τα κράτη-μέλη δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα κονδύλια. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη δεν ήταν σε θέση αυτά τα μη χρησιμοποιηθέντα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν για άλλες δραστηριότητες. Ειδικά οι χώρε βεβαίω που πληρώνουν ήταν ε, πολύ ικανοποιημένε που δεν έπρεπε τελικά να πληρώσουν όσα είχαν υπολογίσει. Εμεί λοιπόν από την πλευρά τη Κομισιόν εδώ είμαστε διατεθειμένοι αυτά τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά να τα χρησιμοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο για να πάνε σε άλλε δραστηριότητε. Αλλά μέχρι στιγμή η διαθεσιμότητα δεν υπήρχε. Το νωρίτερο είναι το 2014 που θα μπορούμε να ξέρουμε πόσα είναι τα κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και ο Ούγγρος συνάδελφος, για, να το, για να το πω, για να το καταλάβει, δεν έχουμε δεσμευμένες πληρωμές, έχουμε δέσμευση υποχρεώσεων. Υπάρχει, υπάρχει διαφορά. Οι υποχρεώσεις είναι υποσχέσεις για το μέλλον για να κατανεμηθούν κάποια χρήματα για προγράμματα που θα εφαρμοστούν στο μέλλον και είδαμε, βρήκαμε μάλλον ένα δίκτυο ασφαλείας, ειδικά για την Ουγγαρία, να δεσμεύσουμε δηλαδή 29% του, των ετήσιων υποχρεώσεων για τη χώρα αυτή, για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε συνέχιση της εφαρμογής των διορθωτικών ταμείων. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε. Δεν θέλω να απογοητεύω τους βουλευτέ το μισό αυτό. Θα μπορούσα να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στους πέντε που έχουν ζητήσει το λόγο, ένα λεπτό καθένα να κάνουν την ερώτησή τους και μετά μια και έξω να απαντήσετε σε όλους. Ωραία. Τέλεια. Ένα λεπτό καθένα. Ζητώ συγγνώμη. Μπορείτε και να παραιτηθείτε άμα θέλετε, αλλά αυτό έχετε. Ένα λεπτό ή τίποτα. Μοζόν πρώτα απ' όλα από την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και την Οικονομική Επιτροπή της Μάλτας, από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Οι πρωτοβουλίες ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων δεν ε, πρέπει να είναι ίδια πολιτική για όλους, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως για μικρές χώρες όπως είναι η Μάλτα. Είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται είναι για τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να επενδύσει. Τώρα όμως διαπιστώνουμε να γίνεται μετακίνηση χρημάτων από την Ευρώπη προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, αυτό που σας είπα πριν και ο ιδιωτικό τομέα να επενδύσει περισσότερο στην Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σίλινα, Λετωνία, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας επενθυμίσω τις προτερότητες που υπενθύμησε ο κύριος Χάν, που είναι επένδυση στην εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εννοείται ότι αυτή είναι δουλειά που επομίζονται κυρίως τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης και τους ζητάω τα διαρθρωτικά κονδύλια να πάνε στην εκπαίδευση. Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους. Αν δούμε όμως τα στατιστικά στοιχεία, 70% των άνεργων δεν έχουν πάει στο πανεπιστήμιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση και πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα προσέοντα τα οποία χρειάζονται οι νέοι όταν ε, βγαίνουν από το γυμνάσιο, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν και στην οικονομία, αλλά πρέπει να κάνουμε και μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως. Σε πολλές ε, χώρες φαίνεται ότι βοηθάει πολύ η επένδυση στην επαγγελματική κατάρτιση. Και μέσω αυτής μπορούμε να στοχεύσουμε τους νέους. Η κυρία Άρτκιν τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινωνικές Υποθέσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω παρακαλώ. Μιλάμε εδώ για την ανεργία των νέων. Ακούσαμε από την Ισπανία τα, τα ποσοστά και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μιλάμε τώρα και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ναι, αλλά αυτό είναι η προσφορά. Για να δούμε και τι είναι η ζήτηση οι χώρες οι οποίες περνάνε από τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, τι γίνεται εκεί. Ε, καταραίει η κατάσταση. Η Επιτροπή λέει ότι αν κάθε μία μικρομεσαία επιχείρηση δημιουργούσε μία θέση απασχόλησης, τελείωσε ενέργεια. Μα δεν υπάρχει όμως η ζήτηση αυτή για να δουλέψει ο κόσμος. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, ότι δεν υπάρχει δουλειά. Έπειτα μιλάμε με στη μοναδική ίσως χώρα η οποία ψηφίζει όπως θέλουμε, τι μας λένε, μας λένε ότι αν συνεχίσετε θα βγείτε από το πρόβλημα. Ναι, η Ιρλανδία τους στήρισε τους κανόνες, η μόνη χώρα ίσως. Ποιος μπορεί να μας εγκινηθεί ότι αν συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες θα λυθούν τα προβλήματά μας. Εμείς φοβάμαι ότι όσο και να τηρήσουμε τους κανόνες δεν θα βγούμε από το πρόβλημα η ε, Ιταλία τώρα. Τελική Βουλή. Κυρία Πόλη Μπορτών, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν εφήγει. Αυτό της σχέσεως με το σύστημα των τραπεζικών πιστώσεων, με τις τράπεζες. Κυρίως από την πλευρά των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σχέση με εκείνη που θα είναι η επόμενη ρύθμιση, η επόμενη νομοθεσία, η επόμενη οδηγία όσον αφορά τη Βασιλεία 3 που από ό,τι φαίνεται θα μπορούσε να θέσει σε δυσχερή θέση κατά πολύ τις μικρές τράπεζες, τις λαϊκές τράπεζες και τις ε, τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες. Οπότε θα προσπαθούμε να βρούμε ενιαίο μέγεθος ρούχου για διαφορετικά σώματα, χωρίς να κάνουμε διαφοροποίηση. Χωρίς να βλέπουμε ποια είναι η θέσεις, ποιες είναι οι απαιτήσει κεφαλαίων από κάθε τράπεζα και αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τον ιστό, τον κοινωνικό ιστό ε, και κυρίως που σε κάποιες περιοχές σε ύφεση ε, αποτελείται το ιστός αυτός από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άσπρης από το Ιστανικό Κοινοβούλιο της Επιτροπής Κοινωνικών, Οικονομικών Υποθέσεων του Ιστανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω συγκεκριμένες σύντομες ερωτήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τα ιδιωτικά ταμεία και την πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειωθεί η γραφειοκρατία όσον αφορά τη βοήθεια που χορηγείται από τα ιδιωτικά ταμεία όπως είπαν ήδη οι Ιρλανδοί συνάδελφοι εκείνοι ε, ε, αυτοί που εκτέλεσαν, υλοποίησαν πιο καλά τα έργα, απορρόφησαν περισσότερους πόρους. Να πω κάτι την οικονομική ανάπτυξη. Εστονία μετά την οικονομική ανάπτυξη η οικονομική μας ανάπτυξη ήταν 8% πέρσι. Έχουμε αποθεματικά. Δεν πήραμε πολλά δάνεια. Καταφέραμε να τα πετύχουμε αυτά μέσω αύξησης των εξαγωγών και πιο βιώσιμης οικονομίας. Ποια είναι η ιδέα που έχω. Ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί της ανταγωνιστικότητας. Να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά και να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι 1% του κοινού ΑΕΠ μα. Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μπορεί να το πετύχουμε τον ιδιωτικό τομέα. Οι αγορέ των εξαγωγών, όσον αφορά τι εξαγωγέ, δείξαν μεγάλο προστατευτισμό. Θα πρέπει επιγραμματικά να απαντήσετε, κύριε Λεβαντόφσκι, είσαστε μόνο σα, αλλά θα πρέπει να απαντήσετε σε 10 ερωτήσει. Ο κ. Λεβαντόφσκι, ευχαριστεί την Πρόεδρο. Τόσο εύκολο, τόσο εύκολο. Α, δεν πρόκειται να σχολιάσω τις παρεμβάσεις με τις οποίες συμφωνώ. Ο ευρωπαϊκός υπολογισμός βεβαίως δεν είναι το υπέροχο όπλο. Δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν είναι πανάκια. Θα μπορούσε όμως να είναι μια χρήσιμη εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της πρόσβασης στην ε, πίστοση ή στο κεφάλαιο που απαιτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούμε να προωθήσουμε ίσω την καλύτερη παιδεία, τη διαβίου, ε, μέσω των προγραμμάτων διαβίου εκμάθησης, ε, το πρόγραμμα έρασμο ή τι ανταλλαγέ και διάφορα προγράμματα για δημιουργία θέσεων που που θα χρηματοδοτηθούν. Δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των χρηματοδοτικών φορέων είπε η κυρία Πόλη Μπορτόνε. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή παίζει ρόλο εποπτείας περισσότερο. Όταν λοιπόν μπείτε εις βάθος, βλέπετε τις αποχρώσεις των προσεγγίσεων όσον αφορά τα διάφορα ιδρύματα μια στάθμιση της προσέγγισης ανάλογα με το μέγεθος του φορέα προς τον οποίο απευθύνονται και των φορέων εκείνων που έχουν συστημική σημασία για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για τον κύριο Άρς, ε, τα διεθντικά ταμεία, ε, το, οι θέσει ορίων, ανωτέρων ορίων, είναι πολύ επώδυνο μέτρο για να συγκρατηθεί ο γενικό ε, προπολογισμό. Ε, συζητάμε κατά πόσο ονομαστικά, το ονομαστικά θα παγώνουμε τα πλαίσια για τη συνοχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι και μαγικό ραβδί τα διεθντικά ταμεία. Για την περίοδο 2007-2013 υπάρχουν κάποιοι πόροι που μπορούσαν να, να προγραμματιστούν. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε, να υποσχεθούμε πολλά. Πρέπει να υπερασπιστούμε την συνοχή στο μέλλον για ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση. Για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 δεν θα πρέπει να καταλήξουμε μόνο με τον προϋπολογισμό για τον αγροτικό τομέα. Πρέπει να τον υπερασπιστούμε τον τομέα τον αγροτικό. Αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε έρευνα και ανάπτυξη που προσβλέπει στο μέλλον. Συνοχή, μεταναστευτική πολιτική διάφορες πολιτικές που υποχρηματοδοτούνται μέχρι τώρα. Με την κυρία Χάρκιν δεν συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε και πρόβλημα του να ανοίξουμε τις αγοράς εργασίας, να τις ξεκλειδώσουμε. Είναι πολύ άκαμπτη η αγορά εργασίας ε, στην Ισπανία. Διατηρεί το, το κατεστημένο και δεν επιτρέπει στου νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Πέρα από τη ζήτηση, που είναι ένα πρόβλημα σε κάποιε χώρες, η απελευθέρωση αγοράς εργασία και η μεταρρύθμιση αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα κράτη-μέλη. Και άλλο ένα σχόλιο. του κυρίου Κλαπισόν τα σχόλια. Υπάρχει ένα στερεότυπο ότι όλοι κόβουν του προπολογισμού και εμείς αυξάνουμε τον προπολογισμό. Αυτό μου λένε συνήθω. 23 εθνικοί προπολογισμοί για το 2012 έχουν αυξηθεί ονομαστικά. 23 από του 27 προπολογισμού. Στου ονομαστικού όρου δεν είναι μεγάλη αύξηση και δεν ταιριάζει πάντα με τον πληθωρισμό. Ονομαστικά όμω είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει την αύξηση του προπολογισμού λόγω κεκτημένων δικαιωμάτων, περασμένων επιδόσεων και το ίδιο ισχύει και για τη Μεγάλη Βρετανία. Ονομαστικά ο προπολογισμό σα αυξάνεται. Αυξήθηκε πέρσι 2% σε ονομαστικού όρου. Από το 2000 μέχρι το 2011 αυξανόταν με μεγαλύτερου ρυθμού από ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό παρά τη διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ενώση που πήγε από 15 σε 27 χώρε. Και πρέπει να μπει και η Κροατία τώρα. Εγώ θέλω να βασίζουμε σε σωστά στατιστικά στοιχεία τις συζητήσεις μας. Και αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη εκτίμηση. Δεν μπορώ να πληρώσω πέρσι πάνω από 10 δις από αξιώσεις από τη συνοχή που έρχονται πολλές χώρες. Συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο που, ποσά που δεν κατεβλήθησαν προς το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια για την Ισπανία, πάνω από 2 δις για την Ιταλία, λόγω ελλείψεως πληρωμών. Στο τέλος δημοσιονομικών προπτικών, όπου έχουμε σώρευση πληρωμών και επιταχύνεται αυτό. Καθυστερούμε στην αρχή, ξεκινάνε προγράμματα και πληρωμές ήταν στο τέλος τώρα, 2012-2013. Λαμβάνοντας υπόψη και το πληθωρισμό, η αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν επιτρέπει να πληρώσουμε αυτά που θα έπρεπε να πληρώσουμε στι χώρε που έχουν προβλήματα όπω είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, να μην αναφέρουμε την Πολωνία. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τώρα. Είναι μια χώρα που είναι σαν ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν απάντησα στι ερωτήσει γιατί με άλλου συμφωνώ. Συμφωνώ με τον κύριο Αρτουή. Μικρό προπολογισμό, 0,2% όπω είπε και ο Χαν όσον αφορά τις επενδύσεις σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. 20-30% των επενδύσεων προέρχεται μεταφορές και 70% των γεωργικών δαπανών στην Ευρώπη έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Σχεδόν ομοσπονδιακή πολιτική. 7% για έρευνα και ανάπτυξη, 93% από εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά στη Γεωργία αντιστρέφεται εντελώ η αναλογία. 70% από τις Βρυξέλλες και μόνο 30% συγχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσά, στους δύο επιτρόπους, ευχαριστώ σε εκείνους που μπόρεσαν να μείνουν μαζί μας μέχρι το τέλος της ανταλλαγής απόψεων. Κατανοούμε ότι υποστηρίζετε την πρόταση μιας ευρωπαϊκής ονοματολογίας που επιτρέπει να συμπεριλάβουμε του εθνικού υπολογισμού στη δυναμική του ευρωπαϊκού υπολογισμού προ εξυπηρέτηση των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Ευχαριστούμε του τρει συζητητέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου διερμηνεί που μα συνόδευσαν μέχρι το τέλο των εργασιών μα. Και πιστεύω ότι ο καθένα θα μπορέσει να συνεχίσει.